επί της αρχής τουλάχιστον να είναι υπέρ μιας ε, τέτοιας ε, πολιτικής. Επίσης θέλω να πω στην Κομισιόν πως ελπίζω πως ε, επιτέλους θα υποβάλει προτάσεις για έναν τέτοιο φόρο, τις οποίες έχουμε ζητήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάρετς έχει το λόγο. Ευχαριστώ.